Και τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Ο οριστικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στις 11 Ιουνίου σύμφωνα με το άρθρο 149 και έχει διανεμηθεί. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Νομική Επιτροπή ενέκρινε τις εξής δύο εκθέσεις για την ασυλία. 891 κάθετος 15 για τον κύριο Φερέιρα, 0192 για τον κύριο Ζιέφκα. Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 8 του κανονισμού του Κοινοβουλίου, αυτές οι εκθέσεις θα ψηφιστούν, θα τεθούν σε ψηφοφορία στην σημερινή διαδικασία ψηφοφοριών. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Κομισιόν σε σχέση με την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 25ης και 26ης Ιουνίου. Η ομάδα των Πρασίνων δήλωσε ότι ο γύρος των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων αντικατασταθεί από μια εις συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι πράσινοι ζητούν να μην μιλήσουν μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί των ομάδων, αλλά να γίνει συζήτηση με συμμετοχή περισσότερων βουλευτών. Κατά συνέπεια, οι προφορικές ερωτήσεις που αφορούν την διαφάνεια για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα μετακινηθούν σε, μετά τις ψηφοφορίες που θα ξεκινήσει αυτή η περίοδο στις 8.30. Αυτή είναι η συνέπεια της ε, πρότασης. Αν αυτή εγκριθεί θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίλιπ Λαμπέρτη για να διατυπώσει το αίτημα της ομάδας του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που παρουσιάσατε την πρότασή μας. Είναι απλή δικαιολογία Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω η ζώνη του ευρώ περνάει αποφασιστικέ στιγμέ σε ό,τι αφορά το μέλλον τη. Θεωρούμε ότι για ένα τέτοιο θέμα τόσο σημαντικό μέσα στα πλαίσια της συνόδου αυτού, αυτής που συνδέεται με το σχέδιο Juncker και με την συζήτηση για το μέλλον της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της θεωρούμε ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη δικαιολογεί ένα ευρύτερο χρόνο. Ξέρω ότι κύριε Βέμπερ πολλές φορές είναι κάπως ασθενικές και άδειε οι σύνοδοι των Βρυξελών, αλλά αυτή τη φορά είναι ακριβώς το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζίμερ ζήτησε το λόγο για να παρέμβει υπέρ της πρότασης Λάμπερτς. Κυρία Τζίμερ. Θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας μου να υποστηρίξω την, άποψη, την πρόταση των Πρασίνων και του Φίλιπ Λάμπερτς είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς λόγω της, της ε, κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ζώνη του ευρώ να μην περιορίσουμε τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σε μια παρέμβαση μόνο των ε, αρχηγών των, κρατών, των ε, κομμάτων για τα προβλήματα αυτά και ιδίω για το θέμα της Ελλάδος χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι ένα δημοκρατικό μήνυμα, ένα μήνυμα ότι λαμβάνομαι υπόψη μας σοβαρά αυτό το πρόβλημα και πρέπει να δώσουμε λοιπόν το λόγο και σε άλλους βουλευτές για να εκφραστούν. Υπάρχει κάποιος που θέλει να παρέμβει εναντίον της πρότασης του κυρίου Λάμπερτ. Όχι κανείς. Θέλετε το λόγο να μιλήσετε κατά. Όχι. Ωραία, λοιπόν τότε ψηφίζουμε την πρόταση του κυρίου Λάμπερτ. Ε, αν εγκριθεί θα γίνει συζήτηση μακρύτερη. Εάν εγκριθεί θα γίνει μακρύτερη συζήτηση, πιο εις βάθος και οι ερωτήσεις θα γίνουν στις 20 και 30. Αν αντιθέτως δεν εγκριθεί η πρόταση του κ. Λάμπερτς, η συζήτηση θα περιοριστεί στις παρεμβάσεις των αρχηγών των ομάδων. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης του κ. Λάμπερτς? Chi è contro? Chi si astiene? È chiaramente Σαφώς απορρίπτεται η πρόταση. Μα είναι προφανέ το αποτέλεσμα. Αν θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, να κάνουμε. Αλλά είναι τόσο προφανέ. Λοιπόν, σα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. La votazione è chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται η πρόταση. Περνάμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη μετά από αυτή την ψηφοφορία που μένει ως είχε. Πρώτο σημείο.